Κοινοβούλιο. Να έχουμε επομένω αυτή την δίωξη, αυτή τη, τη φήμωση για την ε, ε, κατάρριξη τη ελευθερία της γνώμης και αυτό θα πρέπει να μην αποτελέσει προηγούμενο για το μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Γκόλνης, λέει ο πρόεδρο. Σα ενημερώνω ότι τα χθεσινά πρακτικά διατίθενται πρόσωποι τα θέλει και αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Και τώρα έχουμε τις ψηφοφορίες. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Λάινερ που αφορά την εισαγωγή ζών των ζώων αλλά και φρέσκου κρέατος στην κοινότητα. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Σε cierra ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 533 ψήφους υπέρ. Και τώρα πάμε στην ψήφιση της εκθέσεως. Πάνε, πάνε ο πρόεδρος. Ψήφιση της έκθεσης. Okay. Are, you ready? Yes. Okay. Τι είπατε, τι είπατε. Για τρίτη φορά ψήφισε έκθεση ματέρα όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση για την Λιθουανία. Ψηφίζουμε όλο μαζί το κείμενο, ονομαστικά, και εδώ χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Se cierra la votación. Queda aprobado. 558 ψήφοι υπέρ και εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στην έκθεση επίσης κυρίας Ματέρα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, για την ε, Λιθουανία όσον αφορά την βιοτεχνία και βιομηχανία ενδυμάτων ονομαστική ψηφοφορία για όλο το κείμενο. Ψηφίζουμε. Σε cierra la Εγκρίνεται. 562 ψήφοι υπέρ. Και όταν η διαδικασία θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ που αφορά την ετήσια έκθεση του 2009 για την Ευρωζώνη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Bowles για τον ορισμό του Αντιπροέδρου στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έχουμε το σχέδιο απόφαση χωρίς τροπολογίες και θα το ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία όπως προβλέπει το άρθρο 169. Μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται με 488 ψήφους υπέρ. Και τώρα ψήφισε τις εκθέσεις Αγιάλα που αφορά τον ορισμό του κυρίου Μίλαν Μάρτιν Σμιτ ως μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου. Έχει το λόγο η προτείνασα τον κύριο Τσβίγκλ. Κυρία Αγιάλα. Όχι, για να επιταχύνει τη διαδικασία, παρετούμε το δικαιώματο ε, να μιλήσω. Και τώρα, έκθεση για λασέντρο όσον αφορά τον ορισμό του κ. Μίλαν Μαρτίν ω μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. votación. Ψηφίζουμε και εγκρίνεται με 549 ψήφους υπέρ. Και τώρα στη συνέχεια θα ψηφίσουμε τον ορισμό της κυρίας Μπουτμπερ Γκούτε ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Με μυστική ψηφοφορία αρχίζουμε. Σε Πέρας. Εγκρίνεται ορισμός με 545 ψήφους υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση που αφορά την κυρία Κέρστη Καλκιουλάιντ ως μέλος του Ενεργητικού Συνεδρίου, μυστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Σε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κατάληψη αυτή τη θέση με 561 ψήφου υπέρ και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση τη κυρία Αγιάλα που αφορά τον κύριο Ιγκορ Λούντμπορ ω μέλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Σε Ψηφίζουμε, εγκρίνεται. Η πρόταση με 557 ψήφου υπέρ. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση που αφορά τον κύριο Φαζάκα ω μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Σε cierra la votación. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται η πρόταση για τον κύριο Φαζάκας με 348 ψήφους. Και τώρα η πρόταση για τον κύριο Μπάλκο, μέλο του Συνεδρίου Συνεδρίου. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Μη σου, ναι, αλλά φύγει από το χέρι. θα χαθεί, ε. 556 ψήφου υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε την πρώτη προφορά τον κύριο Λουί Γκαλέα ω μέλο του Ενεκτικού Συνεδρίου. Μυστική ψηφοφορία. Σε Πέρα ψηφοφορία. Η πρόταση εγκρίνεται με 553 ψήφου υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση που αφορά την κυρία Κούμπικ για να καταστεί μέλος του ελεκτικού συνεδρίου με μυστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Se cierra votación. El nombramiento queda aprobado con 500. Εγκρίνεται η πρόταση με 568 ψηφού υπέρ και τώρα η πρόταση που αφορά τον κύριο Γιάννη Κίνστ, μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μυστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Άρα, το 1 τρίτο το τελειώσαμε. Ορίστε. Ορίστε. Πέρας. Εγκρίνεται η πρόταση ε, με 558 ψήφους υπέρ και τώρα η πρόταση υποφορά την κυρία Όιν Οσί ως μέλους του Ελληνικού Συνεδρίου. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η πρόταση με 573 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στα νέα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία για την αποστολή τους. Και τώρα, η έκθεση του κυρίου Λάμστορφ που αφορά την σύσταση προς το Συμβούλιο για την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν έχει παρουσιαστεί, δεν έχει προταθεί κάποια ένσταση. Οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται αυτή η σύσταση. Και προχωρούμε για να ψηφίσουμε τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος για την δεύτερη συνάντηση κορυφής της Ευρώπης όσον αφορά τους Ρωμά. Έχουμε σχέδιο ψηφίσματος από 7 πολιτικέ ομάδε. Κυρία Λάμπερτ, κυρία, κυρία Λάμπερτ, συγχωρήστε με, έχετε το λόγο για προφορική τροπολογία. Ναι, Πρόεδρε. Εγώ έχω αυτή την προφορική τροπολογία η οποία θέλω να ονομαστεί στο σώμα του κειμένου 7α νέο. Και νομίζω έχει λάβει το κείμενο και από ό,τι νομίζω συγκεντρώνει τη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων για αυτό το ψήφισμα. Κατά τον τρόπο θα έχουμε αυτό ως συμπλήρωμα της παραγράφου υπαρθμών 7 και σύμφωνα με αυτήν λέει επομένω, για άλλη μια φορά απευθύνω μέχρι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να εκπονήσει μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά την ε, συμπερίληψη, την ένταξη των Ρωμά και κατά αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουν τι διμενεί διακρίσει και την κοινωνικό αποκλεισμό των Ρωμά στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Υπάρχει κάποιο ε, βουλευτή, και συνάδελφο ο οποίο είναι κατά τη ε, τροπολογία Λάμπερτ. Όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η κυρία Ένωστα επίση έχει μια προφορική τροπολογία για την τροπολογία υπαριθμών 1. Κυρία Ένωστα, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ. Έχουμε δύο τροπολογίε προτείνει. Θέλουμε να απαλληφθεί και που λέει The Council and, το Συμβούλιο και. Πρέπει να απαλληθούν αυτές οι λέξεις. Εκεί που λέει θα, ε, καλούμε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν τους αναγκαστικούς επαναπατρισμούς των μειονοτήτων. Μέχρι εκεί που λέει ε, και να έχουν κοινωνική προστασία και απασχόληση μόλις ε, έχουν επιστρέψει. Υπάρχει ένας που έχει ένσταση κατά της τροπολογίας. Ένσταση. Έχουμε πάνω από 40 ενισταμένους, επομένως είναι απαράδεκτη η προφορική τροπολογία τη και τώρα πάμε για την τροπολογία υπαριθμών 1. Τι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριο Σβόμποντα έχει μια προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 18. Κύριε Σβόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ουσιαστικά απορρίψαμε μια τροπολογία η οποία μέσω της αναδιατύπωσής της ε, ξεπερνούσε τα όρια. Υπάρχουν σε ορισμένες χώρες επαναπροωθήσεις Ρωμά και χωρίς να τους δίδεται σε καμία περίπτωση η δυνατότητα να ζήσουν ε, στην χώρα επιστροφής κάτω από συνθήκες ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια έτσι ώστε να, ε, να εκπληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στην περίπτωση κατά την οποία ε, αποδεικνύεται ότι ε, την χάνουν διακρίσεων στην χώρα προς την οποία αποστέλλονται. Έχει κανείς ένσταση επί της ε, προφορικής τροπολογίας Βόμπεντα. Όχι, επομένως ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Se cierra la votación. Πέρας. Εγκρίνεται με 572 ψήφους υπέρ. Και τώρα έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που αφορά την φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων. δυνάμει του άρθρου 151 έχει δει το λόγο ο κύριος Κάσουμαν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εγώ ήμουν αρχικά ο εισηγητής για την απόφαση τη σχετική με τη Frontex και σας τη συστήνω γιατί πράγματι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να ασχοληθούμε με τις παρεμβάσεις ιδιαίτερα στην Νότια Μεσόγειο. Η Επιτροπή μου όμως δεν με στήριξε και γι' αυτό απέσυρα το όνομά μου από την έκθεση αυτή και σας προτείνω να απορρίψετε την έκθεση η οποία είναι μπροστά σας. Απαιτούνται 369 ψήφοι για να γίνει δεκτή, αλλά εγώ προτείνω σαν τέος εισηγητής να απορρίψετε το ψήφισμα το οποίο έχετε μπροστά σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάσμα και τώρα έχει το λόγο η κυρία Μάλστρομ, η Επίτροπος. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Έχετε μπροστά σας ένα σχέδιο ψήφισμα σε ό,τι αφορά τα σύνορα Σέγγεν και σε ό,τι αφορά την εποπτεία των εξωτερικών συνέρων στα πλαίσια των δράσεων της Σέγγεν στη θάλασσα. Πρόκειται για μια απαραίτητη απόφαση η οποία θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη και το Frontex να έχουν πιο αποτελεσματική ε, δίκηση των εξωτερικών συνόρων και όπως ξέρετε θα αυξηθεί η πίεση όπως γίνεται πάντα αυτή την εποχή στη Μεσόγειο. Η πρόταση περιλαμβάνει κάποιες πολύ βασικές αρχές και διευκρινήσεις των κανόνων που θα πρέπει να ισχύουν για παράδειγμα οι έλεγχοι στα σύνορα και περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις ε, προστασίας των ιδιαίτερων ομάδων. Επίσης ειδική αρρωγή για άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και τεχνικές διάσωσης. Πολλοί είχαν ζητήσει από το Κοινοβούλιο να υπάρξουν τέτοιοι κανόνες και τώρα επιπλέον τις έχουμε μπροστά μας. Οι προτάσεις αυτές και οι αλλαγές που προτείνουμε θα μειώσουν τον κίνδυνο για να, χαθ, να χάνονται ζωές στη Μεσόγειο. Το σχέδιο ψηφίσματος αποτελεί καρπό σκληρών διαπραγματεύσεων και συζητήσεων με τα κράτη-μέλη και με εμπειρογνώμονες από τον ΟΗΕ, από τον υποταρμοστή για τους πρόσφυγες και το καθεξής. Θα δώσει στους θεσμούς μας ένα καλύτερο πλαίσιο για την άσκηση σωστής εποπτείας των δράσεων αυτών, όπου έχουν δαπανηθεί ε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για τις νομικές πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 12 έχει χρησιμοποιήσει για βάση γιατί οι κανόνες που αφορούν ε, την παρακολούθηση των συνόρων και όχι τον έλεγχο των συνόρων, όπως ε, λέει η νομική γνωμοδέτηση του Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου εξέτασε διαδοχικές τεχνικές λύσεις προκειμένου καταρχάς να μην ξανανοίξουν οι συζητήσεις για το θέμα αυτό και κατά δεύτερον να υπάρχουν σαφείς κανονισμοί οι οποίοι θα εγκριθούν μέχρι το καλοκαίρι για τις δραστηριότητες του Frontex. Δυστυχώς δεν βρίσκαμε, δεν βρήκαμε άλλες συναλλακτικέ λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να μην απορριφθούν αυτοί οι κανόνες τους οποίους τόσο καιρό περιμέναμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δίνει το λόγο στον κύριο Μπουσούτιλ. Μισό, μισό λεπτό κύριε Μπουσούτιλ, λέει ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. Στα αγγλικά. Δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα αυτό, ξέρετε κύριε Μπουσούτιλ. Έχετε το λόγο. Αλλά μην ανοίξετε συζήτηση. Πρόεδρε, Ακούσαμε δύο μιλητές, ε, ακούσαμε δύο για να απορρευτεί το ψήφισμα. Κανείς όμως δεν μίλησε υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος. Είναι δίκαιο λοιπόν να μιλήσει κάποιος υπέρ του ψηφίσματος. Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε λέω, ένα λεπτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Λίμπε απέρριψε τους κανόνες αυτούς είναι πολύ απλός γιατί η νομική υπηρεσία απεφάνθη δις, όχι μία φορά, δύο φορές, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερεύει τις αρμοδιότητες της ε, υποβάλλοντας αυτή την πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν απορρίψαμε την πρόταση. Θέλουμε σίγουρα του κανόνε αυτού, γιατί και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που επιθυμεί διακαώ να υπάρξουν τέτοιοι κανόνε, αλλά δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερβαίνει τι ε, εξουσίε τη. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την εδώ του ψηφίσματο αυτού. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι κύριε Κάσμαν. Όχι κύριε Κάσμαν, δεν μπορούμε τώρα να ανοίξουμε συζήτηση. Το προανέφερα αυτό. Όχι κύριε Κάσμαν, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Μόνο είναι διαδικαστικό, αλλά διαδικαστικό διαδικαστικό. Έχετε το λόγο. Όσο περισσότερο συζητάτε αυτό το οποίο θέλω να πω, τόσο πιο πολύ χρόνο θέλετε. Απλά θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Αν καταψηφίσετε την πρόταση αυτή, υποστηρίζετε τα μέτρα τα οποία θα επιτρέπουν τις παρεμβάσεις σωτηρίας στη θάλασσα. Αν ψηφίσετε υπέρ, δεν το κάνετε αυτό. Ψηφίζουμε. είναι υπέρ κατά εγκρίνεται θα γίνει η επαλήθευση ψηφίζουμε Σε cierra votación. Πέρα ψηφοφορία. δεν επιτεύχθη η αναγκαία ειδική πλειοψηφία, οπότε απορρίπτεται η πρόταση. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Γεντρεγεύσκα που αφορά τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της χρήσης του 2011. Ψηφίζουμε την τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Σε Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 549 ψήφους υπέρ. Ψηφοφορία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και καταπίπτει η τροπολογία υπαριθμών 3. This has been adopted. No, it's rejected. No, it's acabamos de rechazar la... Πριν από λίγο απορρίφθηκε η τροπολογία υπαριθμών 8. Σύμφωνοι. Επομένως τώρα θα ψηφίσουμε την υπαριθμών 3. Θα την ψηφίσουμε σε δύο τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 3. Ψηφίζουμε. Se cierra la votación. Queda aprobada con 556 votos a favor. Εγκρίνεται με 556 ψήφου υπέρ και τώρα ψήφου το δεύτερο τμήμα. Σε cierra la votación. Πέρας. Το δεύτερο τμήμα της υπαριθμών 3 απορρίπτεται με 371 ψήφους κατά. Τροπολογία υπαριθμών 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα την τροπολογία υπαριθμών 9. Θα ψηφίσουμε ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Σε Πέρας εγκρίνεται με 558 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία υπαριθμών 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 13 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία με 354 ψήφους κατά. Υπερθυμών 14. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές 16. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε Σε Πέρας. εγκρίνεται με 578 ψήφους υπέρ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 18 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε επαλήθευση για την υπαριθμό 18 ψηφίζουμε Se cierra votación. Εγκρίνεται η τροπολογία με 383 ψήφους υπέρ. Παριθμόν 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωση. 19 υπέρ. Votos en contra. Abstenciones rechazadas. Votamos la 20. Votos a favor. Απορρίτατε υπαριθμόν 20 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα την υπαριθμόν 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται υπαριθμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα γίνει η επαλήθευση για την ε, ψήφιση της τροπολογίας 1. Πέρας. Η παριθμόν 1 εγκρίνεται με 374 ψήφους υπέρ. Παράγραφος 67. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Κατά υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 558 ψήφους υπέρ. Είμαστε ευχαριστητές συνεδρία να σας πω ότι μας έχει επισκεφθεί στα πλαίσια των διακοινοβουλευτικών επαφών μία αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο της Τινησίας. Επικεφαλής ο κύριος Ταμπάρκη που είναι ο πρόεδρος τη Επιτροπή των Πολιτικών Υποθέσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Εξωτερικών Σχέσεων για το Κοινοβουλίο τη χώρα. Επομένω, ολόθερμα καλωσορίσατε. Σα ευχόμαστε κύριε Ταμπάρκη και, ε, και εσεί και τα μέλη τη αντιπροσωπεία και θα πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική θεωρούμε την επίσκεψή σα. Είναι η πρώτη επίσκεψη για τελευταία πέντε αιτία εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις της πολιτικές αλλά και οικονομικές της χώρας σας. Είστε ο πρώτος ε, εταίρος μας όσον αφορά τα, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Και υπάρχει μια αντιπροσωπή όσον αφορά τις σχέσεις με το Μαγρέβο, οπότε και αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο οι πολιτικές επαφές θα συζητηθούν τα ζητήματα δημοκρατίας, κράτους ε, δικαίου, οπότε δεν μπορούμε παρά να σας ε, ευχηθούμε καλή διαμονή και καλή δουλειά. Τώρα, θα ψηφίσουμε την έκθεση Triple όσον αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές για τον προπολογισμό της χρήσης 2011. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Στις δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Υπαριθμό 3. Κατά. Υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν τέσσερα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έχουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές, εγκρίνεται Θα ψηφίσουμε την έκθεση Σκότα που αφορά την πολιτική για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα. Υπάρχει κάποια διόρθωση που αφορά όλες τις μεταφράσεις του κειμένου. Ε, τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 411 ψήφους κατά τροπολογία υπαριθμών 3, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 364 ψήφους υπέρ. υπαριθμόν 5 τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 437 ψήφους υπέρ. Έχουμε τον υπαριθμόν 4. Όχι, καταπίπτει. Ναι. Επομένω θα ψηφίσουμε την υπαριθμό 1. Με ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται με 310 ψήφους κατά. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια με την έκθεση Γερέρο όσον αφορά τις επιπτώσεις τη χρηματοπιστωτική κρίσεω, όσον αφορά τι αναπτυσσόμενε χώρε. Έχει το λόγο κύριο Γερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι όταν φτάσουμε στην παράγραφο 31 υπάρχει μια προφορική τροπολογία και σύμφωνα με όσα συμφωνήσαμε θα πρέπει να σας την διαβάσω τώρα ε, εις τα αγγλικά. Θεωρεί επομένω ότι το πιο δόκιμο είναι να διευκολυνθεί. Το κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάποιε συμφωνίε με τι χώρε πιστωτέ, τόσο ώστε να έχουμε ένα μορατόριο προσωρινό όσον αφορά το πάγωμα του χρέου αυτών των ε, φτωχών χωρών, για να μπορέσουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να εφαρμόσουν κάποιε δημοσιονομικέ πολιτικέ για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τι σοβαρέ συνέπειε τη ε, κρίση. Επίση, θα πρέπει να βοηθήσουμε κάποιε άλλε προσπάθειε, ούτω ώστε να έχουμε κάποιο είδου ε, επιδιαιτησία για τον διακονισμό του χρέου και αυτή να είναι με διαδικασίε διάφανες. Θα ευχαριστούμε κύριε κύριε Πάντως, εάν δεν κάνουμε λάθος, αυτή η προφορική τροπολογία αφορά την παράγραφο όχι 31 που είπατε, αλλά την υπαριθμό 34. Γερέρο. Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Είναι το δεύτερο μισό της υπαριθμό 34. Σωστό. Πολύ ωραίο. Τώρα τα πράγματα είναι σαφή, λέει ο πρόεδρος, για να δούμε υπάρχει κάποια ένσταση όσον αφορά την ε, τροπολογία Γερέρο. Την προφορική. Όχι, καλώς. επομένω. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε τη σχετική παράγραφο, θα την ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία του κ. Ιερέρα. Ψήφισε τώρα την παράγραφο υπαριθμών 7, εις δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Το 7, το 7 εις δύο τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ για το πρώτο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα, με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας και εγκρίνεται με 380 ψήφους υπέρ. Πράγμα 22. Ο κύριος Γκέρενς έχει προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωστοποιήσαμε μία προφορική τροπολογία σχετική με την παράγραφο 2. Θυμίζω ότι η παράγραφος 22 έχει σχέση με την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και τη σύνθεση της ομάδας των 20 η οποία δεν περιλαμβάνει κανέναν εκπρόσωπο των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Η προφορική τροπολογία καλύπτει το κενό αυτό και το κείμενο το οποίο προτείνω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται ακριβώς στην έλλειψη αυτή. Πρόεδρος, υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία του κ. Γκέρενς. Επομένως, τότε θα ψηφίσουμε την παράγραφο 22 όπως τροποποιήθηκε προφορά από τον κύριο Γκέρνης ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά θα κάνουμε μια επαλήθευση ψηφίζουμε τώρα ¿eh? Queda aprobado por 282 votos a favor. με 268 ψήφους υπέρ. Και όταν είπε η παράγραφος 23 πει είναι υπέρ. Votos en contra. Abstenciones rechazado. Votamos el apartado 31 en dos 31. Εις δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται θα γίνει επαλήθευση. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της παραγράφου 31. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 287 ψήφους υπέρ. Το δεύτερο τμήμα τώρα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει Τόσο ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ψηφίζουμε. Σε φιέρα βοτασιόν Πέρας, επομένως συγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα με 289 ψήφους υπέρ. Votamos el 34 34 με την προφορική τροπολογία του κύριου Γκερέρο. Τι είπατε κύριε Vous avez την Μπορείτε να του ζητήσετε να κάνουν κάτι για να απελευθερώσουν τον Ταουφίκ Μπεν που ζητάει όλο το κοινοβούλιο την απελευθέρωση του Ταουφίκ Ehm, Του το είπατε εσεί, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ κι εγώ. Σα άκουσα. Πάμε τώρα στην παράγραφο 34 για να ψηφίσουμε την παράγραφο όπω τροποποιήθηκε προφορικά από τον κύριο Γκερέρο. Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα την παράγραφο αυτή. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Από χέρια συγκρίνεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, από χέρια συγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο. Bueno, bien, bien. Vamos a comprobar la segunda... Θα γίνει η επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 34. Ψηφίζουμε. Σε cierra Πέρασε. Está aprobada 300... Εγκρίνεται με 345 ψήφους υπέρ. Και τώρα υπάρχει μόνο 36 δύο τμήματα. Η πρώτη, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Και... Θα κάνουμε παλέψη για το δεύτερο τμήμα της ε, διατάξεως 36. Ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται με 294 ψήφους υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε την παράγραφο 45. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 51. Υπέρ. Κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του κειμένου ψηφίσματος υπέρ το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε επαλήθευση ψηφίζουμε πέρας και τώρα Ατόμη ψηφορία κρίνεται ότι εγκρίνουμε την ε, πρόταση ψηφίσματος με 283 ψήφους υπέρ. a votar el informe Έκθεση Σικλούνα. Ναι, κύριε Σβόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Χαίρομαι για την ψηφοφορία όπως εξελίχθηκε, αλλά ήταν έκθεση πρωτοβουλίας ε, και είχε συμφωνηθεί διαφορετική διαδικασία. Επιτρέπεται σε τέτοιες εκθέσεις να κάνουμε μία και μοναδική ψηφοφορία. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί τελικά θα καταλήξουμε σε όλες τις εκθέσεις πρωτοβουλίας να ψηφίζουμε μονομένα. Θα μπορούσατε να ζητήσετε από την Επιτροπή ΑΦΚΟ να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί να μην καταστρέφουμε την όλη, το όλο νόημα των μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Eh. Ναι. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια σε τμήματα ψηφοφορία. Γιατί ακριβώ αυτό έχουν ζητήσει οι πολιτικέ ομάδε. Εν πάση περιπτώσει, όλα επιδέχονται αναθεώρηση, τροποποίηση ει το μέλλον. Αλλά σήμερα αυτό ισχύει. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Σικλούνα που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κείμενο του 2008. Θα ψηφίσουμε κατευθείαν το σχέδιο του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες, τις ψηφοφορίε. Έχουμε τις κοινέ θέσει του Συμβουλίου ει πρώτη ανάγνωση. Με ε, τις προτάσει τη Επιτροπής σε σχέση με την σύνοδο. Έχουμε τρει μήνε, ούτω ώστε να τοποθετηθούμε και από αύριο αρχίζει να τρέχει αυτή η προθεσμία η τρίμηνη, ούτω ώστε να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο. Τα πρακτικά τη ε, Συνόδου πρόκειται να υποβληθούν προ έγκριση στο Κοινοβούλιο κατά αρχά τη ε, επομένη Συνόδου. Και τα κείμενα των ε, ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν θα τα διαβάσουμε αρμοδίως. Τώρα έχουμε τι δηλώσει τη σχετικέ με την ψηφοφορία. Όσον αφορά την ε, συνάντηση κορυφή για του Ρωμά, έχει τον λόγο κύριο Πάσκα. Ďakujem za slovo, vážený pán e, predsedajúci. E, prijatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom Európskom samite o Rómoch. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή